και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θεωρούνται εγκεκριμένα. Να σας ενημερώσω ότι σήμερα έχουμε την αντιπροσωπεία του ε, Πατριάρχη του Κιέβου και ολόκληρης της Ουκρανίας και την επίσκεψη της ομάδας που τον ακολουθεί. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ και ε, φέρει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της ειρήνης μαζί του. Είναι τιμή να σας φιλοξενούμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μετά την, του, μετά την παρέτηση του Ζαν Φιλίπ Άλπερτ και την ε, χειρία